Ah, where's my button? That one. So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι που μπορώ να σας χαιρετήσω εδώ. Άρχισε η συνεδρίαση. Ταυτόχρονα θα ήθελα να πω την προσοχή στο γεγονός ότι κατόπιν έχουμε ψηφοφορίε. Και βέβαια δεν θα χαρούν οι συνάδελφοι αν καθυστερήσουμε. Και γι' αυτό σας παρακαλώ να τηρήσετε το χρονογόρευση. Δεν θα είμαι πάρα πολύ ε, επίκης. Το πρόσημο σημείο της διάταξης είναι η έκθεση του κυρίου Κάλλος Χωσέη Τούρκα Σανκούλο για εφαρμογή οδηγία για διαχείριση των αποβλήτων. Θα ήθελα αμέσω να δώσω το λόγο για τέσσερα λεπτά στον εισηγητή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψατε μου να αρχίσω για αυτή την ε, έκθεση ευχαριστώντας την Γραμματεία για το έργο που επιτέλησε, τη Γραμματεία της Επιτροπής των Αναφορών την Καρολάιν και τους ε, μου που οι συνεργάτες μου με την ε, βοήθειά τους κατέστησαν εφικτό το να ε, προετοιμαστεί αυτή η έκθεση και σχεδόν επί ένα χρόνο επεξεργαζόμαστε αυτήν την έκθεση όσον αφορά τα απορρίμματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είχαμε διάφορες αναφορές οι οποίες κατήγγυλαν την ε, κακή διαχείριση όσον αφορά ε, το, κάποιες χωματερές όσον αφορά την ε, καταστροφή του περιβάλλοντος και η Επιτροπή των Αναφορών πάντοτε δέστητη σε τέτοια αιτήματα, έκανε κάποιες αποστολές διαπίστωσης, ούτως ώστε να μπορέσουν επί τόπου να, να, να, να διαπιστώσουν ακριβώς τι γίνεται όσον αυτές τις καταγγελίες. Και έτσι φτάσαμε εδώ, ε, στην Ολομέλεια, γιατί είπαμε ότι θα πρέπει να δούμε ε, πώς θα μπορέσουμε να επαγρυπνήσουμε και να δούμε πώς θα εφαρμοστεί ορθά η νομοθεσία από τα κράτη-μέλη. Και όπως έλεγα στην αρχή της παρέμβασης, οι περισσότεροι από τους Ευρωπαίους προσδοκούσαν οι δημόσιες υπηρεσίες να είναι αποτελεσματικές όσον αφορά τα θέματα υγείας, παιδείας, μεταφοράς και ασφάλειας. Παρ' όλα αυτά, το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε ένα σωρό αναφορές, διότι από ό,τι φαίνεται δεν είναι στέσιν οι δημόσιες αρχές, τόσο ώστε με ικανοποιητικό τρόπο να μπορέσουν να ρυθμίσουν το θέμα αυτό των απορριμμάτων και αποβλήτων. Και έχουμε υιοθετήσει ένα σωρό νομοθετικά μέτρα, τα οποία ισχύουν σε όλα τα κρατημέλη και έτσι θέλουμε να μπορέσουμε να έχουμε τις εγγύσεις για να ισχύσει η νομοθεσία και έτσι να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ε, στο ότι σύγχρονος τρόπος ζωής δημιουργεί πάρα πολλά σκουπίδια και στο, στον τόπο δουλειά και από τη βιομηχανία και ακόμα και από τα νοσοκομεία. Οπότε αυτό το οποίο είναι φανερό ότι αν δεν δοθεί προτεραιότητα σε αυτό το πρόβλημα θα έχουμε πολύ αρνητικά αποτελέσματα και όχι μόνο για την υγεία και την ευημερία αλλά ακόμα και για την ίδια την ύπαρξη του πλανήτη. Ανησυχούν επομένω οι τοπικέ κοινότητε και ότι η διαχείριση έχει γίνει ένα σοβαρό πρόβλημα κοινωνικό και πολιτικό και προσδοκούν οι Ευρωπαίοι να επιλύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το πρόβλημα αυτό. Η ανάλυση των πολιτικών που ισχύει στα κρατημένα σε σχέση με αυτό ε, μας έδειξε ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αντιφάσεις και επίσης πάρα πολύ σημαντικές παραλήψεις όσον αφορά την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας η Επιτροπή των Αφορών το 2011, μάλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, ε, είπε και ανακοίνωσε ότι έχουμε 77 παραβιάσει του κοινωτικού δικαίου όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων και τι χωματέρε και είπαν ότι θα πρέπει επομένως ε, να υπολογίσουμε, να συνυπολογίσουμε μάλλον ότι έχουμε 619 παρόμοιε χωματερέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, και επομένως ε, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε περισσότερη ανακύκλωση και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να επιληθεί αυτό το πρόβλημα της διαχείρισης των ε, απορριμμάτων. Έχω υποβάλει σχετικέ προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει να μην ξεχνούμε σε σχέση με αυτό ότι έχουμε μία σειρά από διαδικασίες επί παραδιάση του δικαίου ε, που έγιναν επειδή δεν εφαρμόζεται το κοινωνικό δίκαιο και όμως από πλευρά των ε, αναφερόντων ακόμα πάρα πολλά θα πρέπει να γίνουν όσον αφορά την ε, εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και ακριβώς συνδέεται με το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων οι οδηγίες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και διακόπτει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Ξενοτόμος της Επιτροπής, η κυρία Γεωργίευα έχει το λόγο τώρα για τρία λεπτά. Uh, uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Θα ήθελα εξ ονόματος της ε, βουλευτή της Επιτροπής ε, να συγχαρώ τον εισηγητή για την εξαιρετική έκθεσή του για τη διαχείριση των ε, αποβλήτων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους υπόλοιπους βουλευτές για τις παρεμβάσεις τους σε αυτό τον σημαντικό διάλογο. Καλωσορίζουμε την έκθεση γιατί περιγράφεται η τάξη πραγμάτων σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων και την εφαρμογή της σχετικής οδηγίας στα κράτη-μέλη. Η πλήρης εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας είναι απαραίτητη για ένα υγιές περιβάλλον και για να διαθέτουν του απαιτούμενους πόρους στον τομέα της βιομηχανίας. Μετά την εφαρμογή της οδηγίας βλέπουμε μεγάλες ανισορροπίες ε, στα κράτη-μέλη ως προς τη διαχείριση των αποβλήτων. Κινδυνεύει λοιπόν το περιβάλλον μας, αλλά όχι μόνο, τίθεται εν κινδύνο ολόκληρη η οικονομία και η βιομηχανία δεν μπορεί να αποκομίσει τα ωφέλη της πλήρους εφαρμογής. Κάποια δεδομένα. Πρώτον, δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες ε, λόγω της ελληπέστατης εφαρμογής της οδηγίας. Χάσαμε την ευκαιρία και 72 δις ευρώ είναι το ποσό των ζημιών όπως εκτιμούνται. Δεύτερον, αν διαχειριζόμασταν τα απόβλητα βάση της κείμενη νομοθεσία, θα μπορούσαμε ανάμεσα σε 146 και 244, 264 ε, τόνους συγγνώμη, εκπομπών, θα μπορούσαμε να τους είχαμε αποφύγει. Δηλαδή, 19 ε, με 31% των στόχων που έχουμε θέσει για το περιβάλλον βάση της στρατηγικής της Ευρώπης για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών ε, τίθενται εν κινδύνο χάνονται πάρα πολλές θέσεις εργασίας, ε, θέσεις εργασίας που χρειαζόμαστε δοθεί της ύφεσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα αριθμητικά στοιχεία και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμφωνήσει απολύτως με το συμπέρασμα της έκθεσής σα ότι πρέπει να επισπεύσουμε τη διαδικασία και να εφαρμόσουμε πλήρως ε, την νομοθεσία. Το Κοινοβούλιο καλεί τα κράτη-μέλη να μεταγράψουν εθνική του νομοθεσία τη σχετική οδηγία για την διαχείριση των αποβλήτων αμελητή και να συμμορφωθούν με τις ε, επαιτίες που προβλέπονται συνολική, να υπάρχει συνολική διαχείριση αποβλήτων στις κατάλληλες μονάδες, ε, ε, ούτω ώστε ε, ταχύτατα να εφαρμοστεί η εθνική νομοθεσία που θα μεταγράφει την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Θα συνεχίσουμε να καθοδηγούμε τα κράτη-μέλη για τα, τις πρακτικές επιτυχίες ε, της εφαρμογής ε, της νομοθεσίας. Ε, θα χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τους πόρους μας και θα εστιάσουμε την προσοχή μας στα πλέον προβληματικά κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουμε από κοινού με αυτά τα κράτη-μέλη τις ατέλειες που παρατηρούμε. Επίσης, ενδεχομένως θα ενισχύσουμε τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος πάλι για τις πρακτικές πτυχές της εφαρμογής Εν κατακλείδη θα έλεγα ότι έχουν γίνει κάποιες προσ προσπάθειε για να καλυφθούν οι ανησυχίε που εκφράζει το Κοινοβούλιο μέσα στην έκθεση του. Ταυτόχρονα είμαστε ευγνώμε διότι μας ε, τονώνει τι προσπάθειές μας με την ενέργειά του το Κοινοβούλιο μέσω αυτή τη έκθεση. ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Κατόπιν περνάμε στου συνομιλητές εξ πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Γιάννη, τρία λεπτά από το ΕΛΚ πρώτος. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η έκθεση του κυρίου Ιντουργκάζ αναφέρεται στο πρόβλημα της ε, ε, διαχείρισης των αποβλήτων, ένα θέμα που αποσχολεί πολλούς πολίτες στην Ευρώπη και ευχαριστώ τον συνάδελφο Ιντουργκάζης που μπόρεσε με πολύ καλό τρόπο να προωθήσει αυτή την έκθεση. και το έχει βάλει πραγματικά σε, ένα ουσιαστικό, σε μια ουσιαστική βάση. Υπάρχουν πολλά προβλήματα όσον αφορά τις ιδέες εφαρμογής ε, της νομοθεσίας την αποφυγή, ε, εκμετάλλευση και ε, διαχείριση των αποβλήτων. Η Επιτροπή Αναφορών πολλές φορές ε, με ταξίδια μπόρεσε να δημιουργήσει μια καλή εικόνα της κατάστασης επιτόπου στις διάφορες περιφέρειες λόγω της πλήξης του περιβάλλοντος από το θέμα αυτό πρέπει το πρόβλημα να επιληθεί το γλυγορότερο δυνατόν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλες οι περιφέρειες να εφαρμόσουν σύντομα την σχετική κοινοτική νομοθεσία και να προετοιμάσουν τα απαραίτητα προγράμματα για κάτι τέτοιο. Υπάρχουν οι προτάσεις και θα πρέπει να ακολουθηθούν από τις, από τις ε, χώρες μέλη. Το πρόβλημα βρίσκεται δηλαδή ενώπιον των κρατών μελών. Από την άλλη μεριά βασίζομαι και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα πρέπει έγκαιρα να παρέμβει όταν φανεί ότι η μεταφορά στις περιφερειές ε, δεν γίνεται σωστά και ότι δεν πραγματοποιούνται αυτά που προβλέπει η σχετική κοινοτική νομοθεσία ή όταν βλέπει η Κομισιόν ότι οι περιφερειές δεν μπορούν να προετοιμάσουν τα σχετικά προγράμματα. Επίσης είναι σημαντικό ε, να υπάρχουν και οι σχετικές κυρώσεις. Επίσης ένα σημαντικό ρόλο παίζουν και οι καταναλωτές γιατί εάν δεν γνωρίζουν οι καταναλωτές τι πρέπει να γίνει δύσκολα θα μπορέσουμε να ε, ε, πραγματοποιήσουμε ένα πραγματικό, μια πραγματική ανακύκλωση των ε, αποβλήτων ή μάλλον των πρώτων υλών που περιέχονται σε αυτά. Ε, βέβαια θα πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι τα καλύτερα απόβλητα είναι εκείνοι που δεν δημιουργούν το καθόλου. Αυτό είναι καλό για τους ε, πολίτες, ε, για το περιβάλλον και για τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε. Θα ήθελα λοιπόν κατά κλείδι να πω τι χρειαζόμαστε. Καταρχήν χρειαζόμαστε μια ιδέα της αξιολόγησης και αποφυγής των αποβλήτων. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να προετοιμάσουν οι περιφέρειες. Και συμφωνώ με την Κομισιό ότι αν δεν υπάρχουν σχετικές ιδέες δεν θα χρηματοδοτούν από τι Βρυξέλλε. Σωστό αυτό. Δεύτερον και είναι επίση σημαντικό. Εάν οι υπεύθυνε περιφέρειε δεν είναι σε θέση ή δεν θέλουν να προετοιμάσουν τα προγράμματα αυτά, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αναλάβουν την υποχρέωση αυτή, να βοηθήσουν για να προετοιμαστεί το σχετικό πρόγραμμα. Και αν υπάρχουν και καθυστερήσει χρονικέ, και εδώ είναι η μόνη επίκριση που έχω να κάνω από την Κομισιόν, θα πρέπει η Κομισιόν να βοηθήσει ούτω ώστε τα κρατη να εφαρμόζουν το θέμα αυτό έγκαιρα, ούτω ώστε βουνά αποβλήτων να μην καταστρέφουν το όμορφο τοπίο της Ευρώπης μας. Πρόεδρε, ευχαριστώ, συνάδελφε. Η, για την ομάδα των Σοσιαλιστών, η συνάδελφο Μέρκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, Επίτροπο για τα θετικά που μας είπε. Θα ήθελα να την ευχαριστήσω που συμφωνεί ότι χρειάζεται μια σωστή πολιτική διαχείριση των αποβλήτων. Ακούσαμε στα κράτη-μέλη τους πολίτες να εκφράζονται πάνω στο θέμα αυτό. Στην Ιταλία, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία ακούμε ότι υπάρχουν ακόμα πολλές χωματερές, αλλά δεν υπάρχουν διαπληρίες μόνο από τις χώρες αυτές. Φαίνεται ότι αυτό το πρόβλημα των αποβλήτων υπάρχει παντού και θα πρέπει να λυθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην επιβαρύνει τους πολίτες. Ε, βλέπουμε να λείπει η διαφάνεια. Οι πολίτες θέλουν να ξέρουν τι γίνεται. Θέλουν να ξέρουν πώς αντιδρούν οι αρχές για ένα πρόβλημα που ε, σημειώνουν οι πολίτες. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε ότι θα πρέπει να προσέξει καλύτερα το θέμα η Κομισιόν. Ναι, αλλά δεν τη το ζητάμε αυτό για πρώτη φορά. Πολλές φορές τη ζητήσαμε όχι να πει ότι κάτι πρέπει να γίνει, αλλά πράγματι να κάνει κάτι. Υπάρχουν διατάξεις οι οποίες είναι πολύ καλές μέσα στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε λοιπόν κάποια προγράμματα για την εφαρμογή των ε, διατάξεων που υπάρχουν. Και είπαν ήδη οι συνάδελφοι, θα πρέπει να παρέμβουμε. Χρειαζόμαστε μηδενική ανοχή στην πολιτική μας. Δεν πρέπει να δίνονται πια επιδοτήσεις για να μπορέσει να ασκηθεί πραγματική πίεση στις περιφέρειες και στα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να μπορέσουν πραγματικά να προγραμματοποιήσουν τα διάφορα σχετικά προγράμματα. Εν τελευταία λύση θα πρέπει ίσως να προσφύγει στο δικαστήριο η Κομισιόν κατά των κρατών μελών για να μας πούνε γιατί αδρανούν. Και γι' αυτό έχω τρεις απαιτήσει που υπάρχουν και στην έκθεση. Πρώτον, πολιτική μηδενική ανοχής. Δεύτερον, υποστήριξη κατά την προετοιμασία των προγραμμάτων όταν δεν το καταφέρνει μόνο του το κράτη-μέλη. και σήμερα που είναι η εποχή κρίσης είναι δύσκολο να υπάρχουν ε, το προσωπικό και οι πόροι για κάτι τέτοιο. Και το τρίτο, το σημαντικότερο, είναι η διαφάνεια. Οι πολίτες ζητούν τη διαφάνεια. Χωρίς τη διαφάνεια οι πολίτες θεωρούν ότι βρίσκονται εκτός της διαδικασίας. Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Από πού έρχονται τα απόβλητα αυτά, πού πάνε γίνεται νόμιμα η διαχείρισή τους. Το πρόβλημα είναι μια ευκαιρία. Χρειάζομαστε πρώτες ύλες και εδώ έχουμε μια πηγή πρώτων υλών. Εκεί που υπάρχουν προβλήματα στην Ευρώπη θα πρέπει ακριβώς να δημιουργηθούν οι πιο σύγχρονες περιφέρειες, οι πιο, τα πιο σύγχρονα προγράμματα, γιατί δεν μπορούμε να ε, ακολουθήσουμε διαπολιτική στο μέλλον. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θα ήθελα για την ε, ομάδα των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών δύο λεπτά η κυρία Αλφάνο. Παρακαλώ. Grazie Presidente, tanti auguri per il suo nuovo incarico. Eh, Presidente, io sono molto contenta del fatto che oggi... Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ σωστό το να συζητούμε αυτό το ψήφισμα εδώ ε, στην ε, Ολομέλεια, διότι μια που είναι από εκεί όλων αυτών των ε, αναφορών, οι οποίε έφτασαν στο Κοινοβούλιο όσον αφορά τα απορρίμματα, είναι κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολύ του Ευρωπαίου σε σχέση με τον τρόπο τη διαχείριση. Γιατί είναι θέμα εδώ υγεία, είναι θέμα περιβάλλοντο, είναι θέμα τελικά ακόμα και οικονομία. Οπότε θα πρέπει να επιληθεί αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει τώρα η Ευρώπη και συμφωνώ εν γέννη με το ψήφισμα. Όμω 100% δεν είμαι ικανοποιημένη σε σχέση με κάποιε συγκεκριμένε παραγράφου όπω τα σχετικά με την αποτέφρωση στην κάψη των απορρίτων γιατί και αυτό είναι θέμα ε, υγείας και περιβάλλοντος και δεν ελήφθη όσο θα έπρεπε υπόψη διότι μέχρι και ε, πέρσι εδώ στο ημικύκλιο ακούγαμε ε, τα ίδια όσον αφορά τους σταθμούς πυρηνικής ενέργειας και επομένω σήμερα πώς είναι δυνατόν κάποιος να μιλάει υπέρ των πυρηνικών δεν είναι δυνατόν η πολιτική να μην έχει ένα όραμα ευρύτερο, πιο μακρόπνο ε, γιατί ξέρουμε τι επιδημίες, ε, τι όγκοι ε, δημιουργούνται σε όλους όσους κατοικούν κοντά σε ένα πυρηνικό σταθμό. Επομένως, θα πρέπει να επεραμηθούμε τη ανθρώπινη υγείας, γιατί υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι δημιουργία τη ενέργειας, οπότε θα πρέπει να δούμε και στο θέμα της διαχείρισης των απορρίτων να προχωρήσουμε περισσότερο σε ανακύκλωση. Οι χωματερές είναι μια επιλογή, αλλά δεν είναι πιο καλή. Θα πρέπει επομένω να είναι το Κοινοβούλιο πιο προοδευτικό στι απόψει του. Αυτό προσδοκά ο κόσμο από εμά. Να είμαστε επομένω πιο αυστηροί όσον αφορά και την αποτέφρωση αλλά και τις χωματερές. Επομένω ε, να δείξουμε μηδενική ανοχή. Ευχαριστώ εξ των Κύριε Όκεν, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η έκθεση υποφέρει από παιδικές ασθένειες, θα το έλεγα έτσι. Πολλά μέλη της Επιτροπής μας είναι επιφυλακτικά και δεν θέλουν να απευθύνουν επικρίσεις σε κανέναν. Και θα έπρεπε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι μέσα στην έκθεση. Παρά είναι γενικόλογη η διατύπωση σε σχέση με αυτά που υπόθηκαν στην Επιτροπή Αναφορών στις διάφορες συζητήσεις. Η Επιτροπή Αναφορών ε, δεν μπορεί να λειτουργήσει αισίως ε, αν καθοδηγείται από πολιτικές ε, προθέσεις. Υπήρξε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τον εισηγητή για την έκθεση. Μας άκουσε και κατάφερε να έχει ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα παρά τις παιδικές ασθένειες αυτής ε, της έκθεσης, όπως σας έλεγα στην αρχή. Δεν πιάνουμε τον τάβρο από τα κέρατα. Αυτό είναι το πρόβλημα με την έκθεση. Δεν συνεργάζονται οι περιφέρειες, οι πόλεις μεταξύ τους. Δεν αντλούμε τα διδάγματα από τις επιτυχίες των άλλων. Δεν συμμετέχουν οι πολίτες. Δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε αυτό το πρόβλημα αν δεν εμπλακούν αμεσότερα οι πολίτες. Πολλοί πολίτες στην Ιταλία παραδείγματα παραδείγματα χάρη μας λένε ότι θεωρούνται ως εχθροί σε αυτό το τομέα και είναι πάρα πολύ δυσάρεστη αυτή τους η εμπειρία. Στην ε, Βουλγαρία δε και στην Ισπανία ίσως είναι κάπως καλύτερη η κατάσταση αλλά πραγματικά ο χείριστος μαθητής είναι η Ιταλία. Έχουμε επίσης διάφορες κρίσεις. Καταρχάς μια κρίση ως προς τους πόρους. Ε, θα ήταν ανόητο να ρίξουμε στις χωματερές ε, τους πόρους που έχουμε και όχι να τους ανακυκλώσουμε. Ακόμη ε, πιο ανόητο είναι να αποτεφρώσουμε τους πόρους αυτούς. Αν θέλετε οπωσδήποτε να επιλέξετε την αποτέφρωση. Θα πρέπει να αδειάσουμε τους χήτα, να εφαρμόσουμε σωστά την οδηγία και με ευφυή τρόπο να ανακυκλώσουμε τους πόρους, ε, ούτω ώστε με σύγχρονο τρόπο να εφαρμόσουμε την πολιτική διαχείριση αποβλήτων. Αυτό είναι ο στόχος. Σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Από πλευρά ε, του ECR, κυρία Γκίρλινγκ, τρία λεπτά. Um, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω την έκθεση από πλευράς της ομάδας μου. Ασχολούμαι με το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων στο Κοινοβούλιο επειδή ανήκω στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον όταν διάβασα αυτήν την έκθεση και πραγματικά ε, διαχωρίζεται σε σχέση με προηγούμενες. Ε, δηλαδή ε, δεν υπερασπίζει τα συμφέροντα των ημετέρων, πώς να το πω, και είμαι και επίοικης. Ορισμένοι υπερασπίζουν τα συμφέροντά τους και εμποδίζουν τους άλλους να έχουν μια σφαιρική εικόνα του προβλήματος. Μια τέτοια έκθεση λοιπόν από αυτή την πλευρά είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Αυτό αντικείμενο της έκθεσης ε, αγγίζει όλους τους ανθρώπους που εκπροσωπούμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Ε, όταν εκπροσωπώ την εκλογική μου περιφέρεια, ξέρετε, ε, παρατηρώ ότι οι ψηφοφόροι μου παθιάζονται σπάνια τόσο πολύ για κάποια θέματα όπως για το θέμα της διαχείρισης ε, των αποβλήτων. Και θα κρυθεί λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν δεν τα καταφέρουμε, αν δεν εξασφαλίσουμε την σωστή εφαρμογή της οδηγίας, τότε όλα αυτά τα λόγια που ακούμε εδώ μέσα θα είναι κενά νοήματος. Όλες αυτές οι ιδέες περιέχονται στην πολύτιμη και χρήσιμη αυτή έκθεση. Φυσικά παρατηρούνται με μεγάλες διαφορές ως προς την εθνική διαχείριση ε, του προβλήματος ε, των αποβλήτων. Εγώ όμως καλωσορίζω τις ε, διαφορές αυτές και την έκθεση όπου, τονίζεται αρκούντος ε, η αρχή της επικουρικότητας. Πρόκειται για μια οδηγία πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων και η προκάτοχός μου, η Καρολέν Τζάξον, δεν ξέρω αν τη θυμάμαι, που ήταν η συγγήτρια για την οδηγία πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων. Λοιπόν, μία από, την αρχή, ε, τις αρχές που υποστήριξε περισσότερο είναι η εξή. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν τη μέγιστη δυνατή επικουρικότητα στα πλαίσια όμως δεσμευτικών και δύσκολων στόχων. Σε πρόσφατες συζητήσεις που είχα μαζί της, ε, μου δήλωσε λίγαν απογοητευμένη ε, σε σχέση με την ελευθερία αυτή που έχουν τα κράτη-μέλη, διότι δεν ανταποκρίνονται στους στόχους οι δράσεις ε, των κρατών μέλων παρά την ελευθερία που έχουν. Άρα θα πρέπει να γίνουν πιο αυστηροί οι κανόνες ε, και νομίζω ότι δεν χρειαζόμαστε ένα νέο φάσμα νομοθετημάτων, απλώς χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο που να μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα, αισιότερα. Αυτή είναι η λειτουργία και ενός πλαισίου. Εάν τα κράτη-μέλη λοιπόν δεν εργαστούν μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Σοκαρίστηκα από τον ε, αριθμό των ε, παραβιάσεων ε, που παρατηρήθηκαν από την Επιτροπή Αναφορών και όχι μόνο εγώ αλλά και οι συνάδελφοι. Να προσθέσω και κάτι. Εγώ θα μπορούσα να υπερασπιστώ την πυρηνική ενέργεια όπω και άλλοι, αλλά χρειαζόμαστε σωστή τεχνολογία που θα ελέγχεται αυστηρά. Και το ίδιο ισχύει και για την αποτέφρωση των αποβλήτων. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Επόμενο, εξ ονόματο τη ο κύριος Ενάμιση λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η έκθεση του συναδέλφου Αγκούλο, ο αριθμός και το περιεχόμενο των αναφορών πολιτών και φορέων που ήρθε στην Επιτροπή αποδεικνύουν δύο πράγματα. Πρώτο, ότι το πρόβλημα των αποβλήτων, των απορριμμάτων είναι οξύτατο και φλέγον και δεύτερο, ότι δεν υπάρχουν, με διαβαθμίσεις βεβαίως, ικανοποιητικές επιδόσεις από τα κράτη-μέλη στη διαχείριση των αποβλήτων με προβλήματα στην υγεία και στο περιβάλλον. Ένα σημείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ, όπως το υπογραμμίζει και η έκθεση, ενώ κατά την κοινοτική νομοθεσία η υγειονομική ταφή θεωρείται η εσχάτη λύση, υπάρχουν χώρες όπως η χώρα μου αλλά και άλλες που καθυστερούν στην ανακύκλωση, στην πρόληψη, με συνέπεια να πιέζονται να επεκτείνουν τους υπάρχοντες χώρους ταφής ή να δημιουργούν καινούριου παραβιάζοντας την κοινοτική νομοθεσία, παραβιάζοντας την κοινή λογική, δημιουργώντας οξύτατα προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες, με συνέπεια να έχουμε συγκρούσεις, αλλά και λύσεις επικίνδυνες για το περιβάλλον και για την υγεία. Και το δεύτερο που ήθελα να παρατηρήσω, επικαλούμενο στην έκθεση, αναφερόμενος και στην Επίτροπο, υπάρχουν περιπτώσεις που η Κομισιόν νύπτει τα σχήρα της ή κάνει ή αδιαφορεί για να παρέμβει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Πότε, όταν στην επεξεργασία του σχεδίου για τη διαχείριση των απορριμμάτων στις, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων υπάρχουν πρόδειλα σφάλματα. σε μια τέτοια περίπτωση κυρία επίτροπε πρέπει να παρεμβαίνει η κομισιόν και νομίζω γενικώ κύριε πρόεδρε ότι η έκθεση είναι μια χρήσιμη οδηγία προκειμένου να μας βοηθήσει στη διαχείριση των απορριμμάτων. ευχαριστώ πολύ εκ νόμου του ομάδας του, ο κύριος Ένα μισή λεπτό. Παρακαλώ. Ε, εξ αρχή συγχαίρω τον συνάδελφο τον κύριο Εντουργκάης για την εξαιρετική έκθεση που συνέταξε, την οποία στην Επιτροπή την είχαμε συζητήσει και του είχαμε δώσει τα συγχαρητήριά μα από την πρώτη ανάγνωση. Οι Ευρωπαίοι πολιτέ αναμένουν από τι κρατικέ αρχέ να παρέχουν επαρκεί και αποτελεσματικέ υπηρεσίε ιδιαίτερα στον τομέα των αποβλήτων τα οποία έχουν τεράστια επίδραση και επιβλαβείς επιδράσεις στην υγεία των πολιτών και στο περιβάλλον. από τις επισημάνσεις του οηε τα προβλήματα μέχρι το 2030 της ανθρωπότητος ιεραρχούνται στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, στη μετανάστευση και στα θέματα περιβάλλοντος. Πρέπει λοιπόν, δεν ξέρω αν η ιεράρχηση αυτή είναι σωστή, αλλά πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία σε αυτό οι αναφορές στην επιτροπή αναφορών σχετικά με το θέμα είναι το πιο σύνηθε περιστατικό. συνιστώ λοιπόν όπως σωστά τονίζεται στην έκθεση την εφαρμογή της οδηγίας του 2008 για τα απόβλητα η οποία ορίζει τους κανόνες και την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας προλαμβάνοντας ή και μειώνοντα τι αρνητικέ επιπτώσει τη παραγωγή και τη διαχείριση αποβλήτων. πόροι χώροι πολίτες και όταν λέω πολίτες εννοώ την διαπαιδαγώγηση την εκπαίδευση των πολιτών και διαφάνεια στη διαχείριση των αποβλήτων διότι η διαχείριση των αποβλήτων είναι και ένα μεγάλο οικονομικό γεγονός πρέπει να, να είναι εκείνα τα οποία πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε όλη την ευρώπη. ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο επόμενο ομιλητή, ο κύριο Μέλτσορ, ένα μισή λεπτό. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δύο δισεκατομμύρια τόνοι απόβλητα και από αυτά 40 εκατομμύρια έκτακτα απόβλητα υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, ε, ε, Βλέπουμε ότι ο ρόλος ε, της, ε, της Ευρώπης είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ε, στην Αμερική και άλλες χώρες ε, έχουν προχωρήσει ως περισσότερο. Αλλά εδώ έχουμε πάρα πάρα πολλά προβλήματα. Δεν πρέπει να παραβλέψουμε τις εξελίξεις της ΕΠΑ. Η παρογή ηλεκτρονικών συσκευών ε, στέλνουν τα, τις μη, μη πλέον χρησιμοποιούμενες ε, συσκευές στην Αφρική σαν αναπτυξιακή βοήθεια. Από την άλλη μεριά στέλνουμε εμείς τις πλαστικές ε, μπουκάλες στην Κίνα που χρησιμοποιούνται ούτε ξέρω γιατί. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν έχουμε τόσο πολύ καλή ιδέα ανακύκλωσης. Ε, ένα πολύ μικρό ποσοστό μονάχα ανακυκλώνεται. Το δύσκολο είναι ότι τα απόβλητα μεταφέρονται ανά την Ευρώπη και εναποθέτονται παράνομα. Θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος όσον αφορά τις εξογές των ηλεκτρονικών αποβλήτων και επίσης το θέμα της καταμέτρησης των, ε, του κόστους των μεταφορών αυτών. Επίσης, όσον αφορά επικίνδυνα δηλητηριώδη απόβλητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, δείχνει πάρα πολύ καλή. Θα πρέπει λοιπόν επίσης να δούμε το θέμα των πυρηνικών αποβλήτων και να μην κατασκευάζουμε άλλες πυρηνικέ μονάδες. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Ματσόνη, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον εισηγητή τον κύριο Τουργκάιθ για το έργο του. Αυτή η έκθεση τη πρωτοβουλία ακολούθησε μια απέτηση πολλών Ευρωπαίων πολιτών οι οποίοι υπέβαλαν ένα σωρό αναφορές. Κατήγγυλαν πραγματικά περιστατικά τα οποία ήταν αποκύημα της μη εφαρμογής του κοινωνικού δικαίου. Εδώ είναι θέμα περιβάλλοντος, είναι θέμα διαχείρισης των αποβλήτων. 114 αναφορές έχω μετρήσει σε ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Προέρχονται από 16 διαφορετικές χώρες. Και σε μερικές χώρες τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, σε Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία. Συνήθως αυτό το οποίο ζήτουσαν οι Ευρωπαίοι αφορούσε το ότι δεν έγιναν αυτά τα οποία θα έπρεπε όσο αφορά τη διαχείριση αλλά και την αποτέφρωση των αποβλήτων. δεν εφαρμόστηκαν επομένω οι νέε τεχνολογίε που προβλέπονται για τέτοιε περιπτώσει. Πρόκειται για έναν κλάδο πολύ σημαντικό. Τόσο το μάλλον καθώ περνούμε μια συγκυρία σοβαρή χρηματοπιστωτικής κρίση. Έχουμε παραλάβει πολλές φορές και προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία και εκείνη το ισχυρίζεται ότι θα πρέπει να γίνει διαφορετική χρήση των ε, αποβλήτων και αυτό θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση 70 εκατομμυρίων ευρώ επίσης όμως θα οδηγήσει και σε δημιουργία πολλών χιλιάδων θέσεων εργασίας. Επομένως έτσι θα βοηθήσουμε και, και τον πλήρων αλλά και το περιβάλλον. Ευχαριστώ. Η κυρία Παλαδέλη, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, και εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον συνάδελφο κύριο Ιτουργκάης για την πραγματικά πάρα πολύ ε, προσεκτική, σοβαρή, αντικειμενική και εν τέλει διδακτική προσέγγιση σε ένα θέμα τόσο σημαντικό όπως αυτό το οποίο βιώνει η Ευρώπη των τελευταίων ε, χρόνων. Ε, θεωρώ ότι οι υποδείξεις αυτής της έκθεσης, σε ορισμένα τουλάχιστον σημεία, μπορεί να επιτρέψουν στην Επιτροπή αλλά και στα κράτη-μέλη να προσαρμόσουν τις πολιτικές τους προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που άνισα βέβαια κατανεμημένο στα διάφορα κράτη τη ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργεί, ε, παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Θεωρώ βασική υποχρέωση των κρατών μελών να ενημερώσουν τους πολίτες τους. Όχι μόνο στα σχολεία, αλλά και να, αποκαταστήσουν την σχέση εμπιστοσύνης για μια υπόθεση που τους αφορά όλου. Ε, όλους. Θεωρώ αυτονόητο ότι στις μετρήσεις για παραβιάσεις περιβαλλοντολογικές πρέπει να έχουμε δεδομένα πιο αντικειμενικά. θεωρώ σημαντική την διασυνοριακή συνεργασία και παραμένω ε, ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Μάνερ, ένα, μισή λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα, Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Ιτουργκάη, τον εισηγητή μας. Είναι ε, εξαιρετική η έκθεση που υπέβαλε. Από το 2004 έως το 2010 η Επιτροπή Αναφορών εξέτασε 114 ε, αναφορές πολιτών σχετικά με διαδικασίες ε, που άπτονται της νομοθεσίας διαχείρισης των αποβλήτων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα θέμα, μια πηγή μεγάλης ανησυχίας ε, για τους πολίτες. Ε, σημειώνονται μεγάλες διαφορές ως προς την εφαρμογή σε επίπεδο κράτους μέλους ε, της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Θα πρέπει να αναλυφθεί ταχύτατα δράση, ώστε να εφαρμοστεί οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα. Μόνο έξι κράτη-μέλη έχουν κατορθώσει να εφαρμόσουν εμπρόθεσμα την οδηγία πλαίσιο. Ας μην ξεχνούμε ότι τα απόβλητα συνιστούν πόρους και θα μπορούσαμε να λειτουργούμε πιο αποτελεσματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μια ορθότερη πολιτική διαχείριση. Ευχαριστώ. Μας χάρισε 30 δευτερόλεπτα η κυρία ε, Μάνερ. Η κυρία Μιράντα, ένα λεπτό έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια για την ε, έκθεσή σας, ε, κύριε Τουργκάης. Ε, μέσα στη χώρα μου, στην περιοχή μου, στη Γαλλικία, δεν εφαρμόζεται σωστά η πολιτική για την συλλογή, διαχείριση, διάθεση των αποβλήτων, όπως λέτε ε, στο σημείο 12 της έκθεσής σας. 42% ε, των αποβλήτων μόνο διατίθεται. Προβλέπετε μία νέα χωματερία από την κυβέρνηση και ακολουθείτε μία ηγεμονική, μία κατασταλτική πολιτική για, τους, ε, για τα απόβλητα. Ε, ε, τρία εκατομμύρια άνθρωποι δεν μπορούν ναι, ναι, να υποφεληθούν ναι, από αυτούς ε, τους πόρους διότι έχει επιλέξει η πολιτική να αποτεφρώσει το ίμιση των αποβλήτων. Επίσης, στα σημεία 16 και 18 της ε, έκθεσης ε, δεν αναφέρεστε στην έλλειψη σωστής ενημέρωσης των πολιτών σε σχέση με τις ε, μονάδες αποτέφρωσης. Εγώ θα ζητήσω να εφαρμοστεί σωστά η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για, τις, για τα απόβλητα και θα ήθελα να τονίσω και πάλι ότι η έκθεσή σας υποστηρίζει την τοπική κυβέρνηση της Γαλλικίας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αγκουράκης, ένα λεπτό κύριε πρόεδρε η έκθεση ενώ περιγράφει τα περιβαλλοντολογικά εγκλήματα που συντελούνται στην διαχείριση αποβλήτων και τις καταστροφικές για το περιβάλλον πρακτικές υιοθετεί όλους τους παράγοντες που τα εκτρέφουν. αντί να προτείνει μέτρα ενάντια στην ασίδωτη ρήπανση από το μεγάλο κεφάλαιο διαφημίζει ανοιχτά την καταστροφική δράση των ομοπολιών του κλάδου χειροκροτεί την οδηγία 2008 χιλιάδες η οποία αναβαθμίζει την ενεργειακή καύση που καταστρέφει το περιβάλλον και θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία πολλαπλασιάζοντας όμως τα καπιταλιστικά κέρδη. η ίδια οδηγία νομιμοποιεί την ασυδοσία του βιομηχανικού κεφαλαίου στη ρήπανση καθώς επιτρέπει την, ανάμειξη επικίνδυνων με μη επικίνδυνα απόβλητα. αναφέρεται η έκθεση στο ρόλο του οργανωμένου εγκλήματος Συνάδελφε, με συγχωρείτε κύριε Συνάδελφε, το λίγο πιο αργά παρακαλώ. Λίγο πιο αργά, γιατί αλλιώς δεν μπορείτε να μεταφραστείτε. Απ' την αρχή δηλαδή να αρχίσω. <laughs> όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Αναφέρεται η έκθεση στο ρόλο του οργανωμένου εγκλήματος στη δημιουργία περιβαλλοντικών κινδύνων για να κρύψει το πραγματικό ε, ταξικό έγκλημα σε βάρος του περιβάλλοντο που διαπράττουν τα μονοπόλια ε, τα όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσει των κρατών μελών. Στην Ελλάδα, στην Αργολίδα και σε πολλέ άλλε περιοχέ, στην Κρήτη παραδείγματο χάρη, η υγεία των εργαζομένων βρίσκεται σε διαρκή κίνδυνο από τι χωματερέ ακόμα και τοξικών λιμάτων που λειτουργούν δίπλα στα σπίτια του. Λύση για μας, για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα, είναι η ανατροπή τη ε, πολιτικής της Ευρωπαϊκής έτσι ε, ώστε να διασφαλίζεται η υγεία ε, των εργαζομένων και η προστασία του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε. Ο κύριος Μπογκέτσια, ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρόκειται για κάποια έκθεση πάρα πολύ καλά ε, εξισορροπημένη και που αναφέρεται στον ε, σημαντικό αυτόν ρόλο που πρέπει να αναλάβουν τα κράτη-μέλη για αυτό το πρόβλημα ε, και βέβαια ε, και σε αυτή την περίπτωση έχουμε μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων ακόμη και μέσα στη δική μου χώρα έχουμε δύο ταχύτητες διότι έχουμε α, κάποιους δήμους και κοινότητες όπου πραγματικά είναι ντροπή αυτό το οποίο γίνεται στην ε, αυτό που γίνεται στη χώρα μας με τα, ε, απορρίμματα. Από την άλλη μεριά βέβαια υπάρχουν και ε, κάποια, κάποιους δήμους και κοινότητες οι οποίες κάνουν αυτό το οποίο πρέπει. Ε, ας πούμε στην Λομβαρδία έχουμε εκεί κάποιου δήμου και κοινότητε που κάνουν αυτό το οποίο πρέπει. Εκεί έχουμε μια σόφρονα αντιμετώπιση του προβλήματος των απορριμμάτων. Οπότε θα πρέπει να δούμε το πώς θα καλύψουμε τις αναφορές που έχουν κατατεθεί αυτές τις καταγγελίες και ε, πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό το οποίο είναι και κάτι το οποίο στέφτει κατά του τουρισμού ε, είναι τελικά μια απειλή και για την υγεία. Κύριε Μπογκέτσο, έχουμε μια μπλε κάρτα από την αλφα Αλφάνο. Θέλετε να δεχτείτε την ερώτηση. Παρακαλώ κύριε Αλφάνο. Ε, credo sia l'ennesima νομίζω ότι για πολλωστή φορά αναφέρεται στην περιοχή που ονομάζει Παδανία ο κ. Μπορκέτσιο. Αυτό είναι επιστημονική φαντασία. Υπάρχει μόνο στα, στα παραμύθια. Μίλησε βέβαια και για την Νάπολη, για την Καμπανία, ε, μίλησε για περιοχές που δική κεντροδεξιά, αλλά παρακαλώ, όταν μιλάτε για Ιταλία, να μας πείτε πού βρίσκεται αυτή η περιοχή, μάλλον βρίσκεται μόνο στα όνειρά σας, στη φαντασία σα Πηγαίνετε και διαβάστε, λέει ο κ. Μποργέτσιο, να βρείτε πού βρίσκεται. Έχω εδώ πέρα ένα επίσημο έγγραφο το οποίο αναφέρεται στην κυβέρνηση της Παδανίας. Ξέρω ότι είναι μακριά από εκεί που μένετε της παδανια ξερω οτι ειναι μακρια απο εκει που μενετε εσεις όμως έχουμε ε, και αυτοκινητοδρόμους που ονομάζονται ε, αυτοκινητοδρόμοι της Παδανίας, οπότε πρόκειται για την χώρα των Παδανών, που όντως είναι οραματιστές. Ευχαριστώ για διευκρίνηση αυτή. Επί της ουσίας της εκθεσής μας, ο κύριος Μπουλόν, δύο λεπτά. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Ιτρουγκάη στον εισηγητή για την ποιότητα των εργασιών του, για τις ε, ατέρμονες διαπραγματεύσεις που έπρεπε να κάνει και για την υπομονή που έδειξε. Φτάνουμε λοιπόν και στην ψηφοφορία της ε, τόσο σημαντικής έκθεση, σημαντικής, ε, διότι παρουσία της Επιτροπής και του Συμβουλίου εκφράζουμε τις ανησυχίες των πολιτών μέσα από αυτή την έκθεση. Να λοιπόν, αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα της Επιτροπής των Αναφορών στην Ευρώπη. Ε, παρατηρείται ότι μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες των πολιτών και φαίνεται αυτό από τις αναφορές, είναι η διαχείριση των αποβλήτων. Καταναλώνουμε αλόγιστα και τώρα συνειδητοποιούμε ε, ότι δεν θα πρέπει απλώς να πετάμε αυτό που δεν χρησιμοποιούμε. Θα πρέπει λοιπόν να ενημερωθούν οι πολίτες ε, και ε, να ευαισθητοποιήσουμε τα κράτη-μέλη. Είναι ανησυχητικό που φαίνεται ότι δεν καταφέρνουν να ελέγξουν τα κράτη-μέλη την κατάσταση. Εμπρόθεσμα μόνο έξι κράτη-μέλη εφήρμοσαν την οδηγία πλαίσιο. Ο αριθμός των καταγγελιών για αυτό το θέμα καταδεικνύει καταδεικνύει την έλλειψη ενίοτε της ε, διαφάνειας ε, ως προς ε, τους χώρους υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων. 75 δις ευρώ αυτή είναι η αγορά των αποβλήτων. Κατα... Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλά συμφέροντα. Θα πρέπει λοιπόν να αυξήσουμε τις κυρώσεις κατά αυτών που εκμεταλλεύονται τις δημόσιες εταιρείες για να πλουτίσουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διαδραματίσει το ρόλο της, να παρακολουθεί τη σωστή εφαρμογή, τις οδηγίες για τη διαχείριση των αποβλήτων. Θα πρέπει επίση να είμαστε αξιόπιστοι πέρα από το να προβάλλουμε το πρόβλημα. Αν συνεχίσουμε να παίζουμε αυτό το παιχνίδι, θα χάνουμε χρόνο και χρήματα για τι επαληθεύσει και κόντρα επαληθεύσει, ε, που δυστυχώ μπορεί να διαρκέσουν και χρόνια. Α ακούσουμε το μήνυμα ε, των, ε, αυτών που υπέβαλαν τι καταγγελίε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Ο Ρίβιο και έχει μια μπλε κάρτα. Δεχόσαστε ερώτηση. Επαναλαμβάνω. Ο συνάδελφο του και έχει σηκώσει μια πλεκάτα. Δεχόσαστε μια ερώτηση. Παρακαλώ. Ναι, σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ρωτήσω τον συνάδελφο Μπουλόν το εξή. Πώ φαντάζεται ότι αυτή η αλυσίδα των αποβλήτων που είναι μια αλυσίδα πρώτων υλών θα μπορέσει στο μέλλον να μετατραπεί σε μια ε, αλυσίδα ωφελίας πρώτων υλών. Πιστεύετε ότι το σχετικό ερευνητικό πρόγραμμα θα μπορέσει να βοηθήσει να εκμεταλλευτούμε σωστά αυτές τις πρώτες ύλες. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπουλό, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Euh, Όπως διατυπώσατε το ερώτημα. Ναι, έχουμε ήδη μιλήσει για την διαλογή των αποβλήτων. Δεν έχω κάτι να προσθέσω σε σχέση με αυτή την ερώτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στον Αλφα Σπυρίλο, ένα λεπτό παρακαλώ. Έχουμε, κύριε Πρόεδρε, εκατοντάδε τέτοιων αναφορών που προέρχονται από πολλές χώρε τη Ένωση. Αυτό μας δείχνει πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα αυτό. Η έκθεση του Γκάιτ τονίζει ιδιαίτερα το θέμα της καταστροφής των παρανόμων απορριμμάτων. Έχουμε πρόβλημα τέτοιο και στην δική μας περιοχή. Έχουμε επίση και πυρηνικά αποβλήτα στην ε, Ιταλία. Θα πρέπει επομένω να δούμε πώ θα ασκηθεί κάποιος έλεγχος ε, όσον αφορά τι εγκαταστάσει των χωματερών. Θα πρέπει να εφαρμόζεται η κοινωτική νομοθεσία. Δεν την εφαρμόζει ούτε η Ιταλία όπω και άλλε χώρε. Και έχουμε επομένω, διακίνηση απορριμμάτων παράνομη. Και αυτό είναι διασυνοριακό πρόβλημα και θα πρέπει επομένως να βρίσκεται δεν η Ευρώπη να λύσει το εν λόγω πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ συνάδελφε. Η κυρία Σάρβα, ένα λεπτό έχει το λόγο. Πρόεδρε, μέσα σε αυτή την ε, έκθεση αναφέρονται 115 καταγγελίες από 15 κράτη-μέλη. Ο πολίτες ε, καταγγέλνουν την πλημμύλη εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα. Είναι όμως μόνο η κορυφή του παγόβουνου και το γνωρίζουμε όλοι. Υπάρχουν ε, περιπτώσεις ε, στην ε, Ρουμανία που ενισχύουν αυτή τη θέση. Περισσότερες κυβερνήσεις αδυνατούν να εφαρμόσουν αυτήν την κρίσιμη για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον οδηγία πλαίσιο. Επίση υπάρχει το θέμα των αποβλήτων της εξορυκτική βιομηχανίας που είναι ιδιαίτερα ε, ανησυχητικό. Εσχάτω, εξέφρασα την ανησυχία μου στο Κοινοβουλίο απευθυνόμενη και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία με ενημέρωσε ότι η οδηγία για τα απόβλητα της εξορυκτική βιομηχανίας επαρκεί ώστε να προστατεύσουμε τον περιβάλλον ε, ακόμη και ε, κατά την, στην περίπτωση επικινδύνων ουσιών. Ε, Βεβαίω, αν δεν είναι ορθή η εφαρμογή αυτή τη οδηγία, όπω και η οδηγία για τη διαχείριση των αποβλήτων, αποκλείεται να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Έχουμε εξαντλήσει τώρα τον κατάλογο των ομιλητών. Περνάμε στη διαδικασία του Έχουμε περισσότερου ομιλητέ από τη χρόνο. Γι' αυτό θα ήθελα να δώσω το λόγο σε εκείνους που ήταν εξ αρχής ε, παρόντες στην ε, συζήτηση αυτή. Κάποια μέθοδος πρέπει να υπάρχει για την επιλογή. Λοιπόν, ένα λεπτό. Η κυρία Μακίνες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά που έχει κάνει για αυτή την έκθεση για τους πολίτες, πολυάρθμους πολίτες που κατέθεσαν τις καταγγελίες. Ε, θα έλεγα ότι υπάρχουν και άλλοι τόσοι που δεν γνωρίζουν το πρόβλημα. Η ευαισθητοποίηση του κοινού πρέπει να ενισχυθεί, να ενημερωθεί το κοινό για τη διαχείριση των αποβλήτων ε, και στο σπίτι και στο χώρο εργασίας. Ε, υπολείπεται μεγάλο έργο από αυτή την άποψη. Αν ε, υποχρεώνονταν οι πολίτες να επισκεφθούν ε, ε, πλημερώς λειτουργούσες χωματερές, Καταλαβαίνουν, ότι θα άλλαζαν την άποψή τους σχετικά με τα απόβλητα. Στην περιοχή μου υπάρχει μια παλιά χωματερή που δημιουργεί σοβαρότατα περιβαλλοντικά προβλήματα και δημιουργεί και για τους περικούς σοβαρά προβλήματα. Θα ήθελα να αναφερθώ στην παράνομη ε, δραστηριότητα που ε, περιβάλλει αυτό το θέμα της διαχείρισης ε, των αποβλήτων. Ευχαριστούμε κυρία Τικάου τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλε αυτέ οι αναφορέ που κατετέθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αποτέλεσμα τη ε, μη εφαρμογή τη κοινωτική νομοθεσία. Ούτε έγινε κανένα είδου διαβούλευση και δείχνει το πόσο ο κόσμο έχει πανικοβληθεί όσον αφορά την κατάσταση για τα απορρίμματα. που θα πρέπει να γίνει η σχετική επένδυση, θα πρέπει να έχουμε καινούργιε στρατηγικέ και θα πρέπει να υπάρχει και κατάλληλη υποδομή και κατάλληλο εξοπλισμό αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βοηθήσει προ τούτο τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει επίση να βρει κάποιου χρηματοδοτικού μηχανισμού. Θα πρέπει να καθοδηγήσει, να δώσει καθεντήρε γραμμέ όσον αφορά αυτέ όλε τι ε, χωματερέ. Κυρίω θα πρέπει να προσέξουμε τι γίνεται για εκεί που έχουμε κοντά σχολεία, νοσοκομεία, γενικά κατοικημένου ε, χώρου. Ε, είναι απειλή αυτό για την υγεία και για το νερό. Θα πρέπει επομένω να γίνει μια δημόσια συζήτηση, διαβούλευση, οπότε θα πρέπει να στηρίξουμε τις τοπικές αρχές, ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν τις άριστες πρακτικές για αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Ο συνάδελφος έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ υποστηρίζω τις ιδέες αυτές που εξεφράστηκαν στην έκθεση του κυρίου Τουρκάης. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι θα πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη σημασία στο θέμα των οργανικών αποβλήτων, ιδίως εκείνης τι περιφέρειες που έχουν ε, πολύ ενεργή γεωργία γιατί αυτά τα οργανικά αποβλήτα χρησιμοποιούνται για καύση συνήθως Πράγμα που σημαίνει όμως ότι έχουμε τεράστιες απώλειες. Αν χρησιμοποιούσαμε τα απόβλητα αυτά με καλύτερο τρόπο θα μπορούσαμε να τα εκμεταλλευτούμε και να έχουμε θετικά αποτελέσματα της αναγκύκλωσης. Ίσως από το, 12 πυλο... το δεύτερο πυλώνα μπορεί η Κομισιόν να επιδοτήσει κάποια τέτοια προσπάθεια. Ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό τώρα. Κύριος Πάσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα. Και γι' αυτό θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει κάποιες σχετικές οδηγίες και να τις στηρίσουν τα κράτη-μέλη. Αρχάς του περασμένου έτους είχατε εκείνη την έκθεση όπου καταγγείλατε τα κράτη-μέλη που δεν έλαβαν υπόψη το περιβάλλον όσον αφορά διαχείριση των αποβλήτων. Και έχουμε ένα σωρό περιπτώσεις κατά τις οποίες εκατοντάδες παράνομες ε, χωματερές υπάρχουν. Θα πρέπει να προσπαθήσετε περισσότερο σε αυτό το μέτωπο. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την επεξεργασία των αποβλήτων, γιατί θα μπορούσε αυτό να αποβεί ε, μια οικονομική δραστηριότητα πάρα πολύ επικερδή. Να κάνουμε κύκλο περισσότερο, να καταβάλουμε περισσότερη προσπάθεια και πιο αποτελεσματικού μηχανισμού για τα σκουπίδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφε. Σα είχα πει ότι δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε το λόγο σε όλου. Γι' αυτό ο τελευταίο ομιλητή του ΚΑΣΤΙΑΗ είναι ο Σνόλφο Σικέρσκι.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 Ε, οι παράνομες χωματερές και αποτεφρωτήρες ε, είναι ένα συχνό πρόβλημα για τη χώρα μας. Ε, συνιστά αυτό κίνδυνο για το περιβάλλον και για τη δημόσια υγεία και συνιστά κατασπατάληση χρημάτων διότι δεν ανακτούμε πολύτιμους πόρους από αυτά τα απόβλητα. Χρειάζονται λοιπόν ενισχυμένες προσπάθειες, κυρίως στην Ήπεθρο, για την ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς τις ευκαιρίες αξιοποίησης που παρουσιάζει μια ε, καλή διαχείριση των αποβλήτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο Επιπρόσθετα χρειάζονται σαφείς προσβάσιμες πληροφορίες ε, για τους ε, καταναλωτές, ε, όχι μόνο για την διαλογή στην πηγή, αλλά και για ολόκληρο τον κύκλο της ζωής αυτών των αποβλήτων. Μία ορθή διαχείριση συνεπάγεται σοβαρότητες επενδύσεις από πλευράς διαφόρων κρατών μελών ε, θα πρέπει να αναδειχθεί σε προτεραιότητα το θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να, να συντρέξει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Θα δίνω το λόγο στην κυρία Γεωργίευα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πραγματικά είμαι ειλικρινά ευγνώμων προς τους βουλευτές του Κοινοβουλίου, διότι βλέπω από τις παρεμβάσεις τους ε, που απηχούν τις ανησυχίες των πολιτών ότι ενδιαφέρονται για το θέμα. Διάφορες παρατηρήσεις. Πρώτον, η ψηστή προτεραιότητα για μας είναι προ... να έχουμε σωστό το κύκλο διαχείριση των αποβλημάτων, δηλαδή ε, διάθεση, διαλογή στην πηγή, ε, διαχείριση και ως έσχατη λύση να μεταφερθούν σε χωματερές τα ε, υπολοιπόμενα απόβλητα μετά από εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Πώς, με ποιο τρόπο μπορούμε να συντρέξουμε τα κράτη-μέλη, καλύτερη καθοδήγηση, ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών, αλλά όχι μόνο, ελέγχοντας τα εθνικά σχέδια διαχείρισης, ώστε να διασφαλίσουμε ότι είναι τα πρόσφορα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Για τα 10 κράτη-μέλη που έχουν <coughs> σοβαρότερα προβλήματα, προτιθέμεθα να ε, διοργανώσουμε μεμονωμένες συσκέψεις για να επισπευθεί η δράση στα συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Ε, προφανώς όταν είναι ατελής, ελλειπής η δράση και κάθε φορά που θα το διαπιστώνουμε στο μέλλον δεν θα διστάσουμε, θα κινήσουμε διαδικασίες επιπαραβάσει παραβάση, ε, ούτως ή άλλω, υπάρχουν δεκάδες ε, υποθέσεις ε, που εκκρεμούν στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας. Ένα τρίτο των περιπτώσεων σχετίζονται με παραβάσεις σε σχέση με την ε, πολιτική διαχείριση ε, των αποβλήτων. Όχι μόνο πρέπει να κάνουμε αυτά που πρέπει στα κράτη-μέλη, αλλά θα πρέπει να δώσουμε και το παράδειγμα για τις ε, αναπτυσσόμενες χώρες, διότι αυτά που συμβαίνουν σε άλλες χώρες επηρεάζουν ούτως ή άλλως την κατάσταση του πλανήτη. Θα συμφωνήσω δε με συναδέλφους ότι ε, σε αυτούς τους ε, χαλεπούς ε, καιρούς από οικονομικής πλευράς είναι στην ευκαιρία εκμετάλλευση, αξιοποίηση των πόρων αυτών των αποβλήτων. Δεν πρέπει λοιπόν να χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Ε, υπήρξε και ένα συγκεκριμένο ερώτημα για τα απόβλητα της εξορρυκτικής ε, βιομηχανίας ε, μετά το ατύχημα βιομάρε και την έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής. Καταλήξαμε στην πλέον αυστηρή οδηγία στον κόσμο, από ό,τι ξέρω, για αυτά τα απόβλητα και είμαστε σε στενή συνεργασία με διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ρουμανία, ούτως ώστε να εφαρμοστεί ορθά η οδηγία. Ε, μία τελευταία παρατήρηση. Συγγνώμη που υπερβαίνω το χρόνο μου. Θα ήθελα να πω κάτι για την ε, ευαισθητοποίηση του κοινού. Εγώ, ξέρετε, ασχολήθηκα με τα θέματα περιβάλλοντος ε, και στην προηγούμενη επαγγελματική μου σταδιοδρομία, διότι ε, ε, αρρώστησε ένα μέλος της οικογένειας μου λόγω της μόλυνσης των υπογείων υδάτων. Υπέστη ανεπανόρθωτες ζημιές και γι' αυτό με ενδιαφέρει τόσο πολύ το θέμα και θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους. Σας ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Και αν μην ξεχνάμε ότι αυτό πρόκειται για μια εκθέση αυναυτή αναφορών, ήταν πάρα πολύ σημαντικό που αναφερθήκατε και το θέμα του κοινού. Ε, τέλος έχουμε τον εισηγητή, κύριο Ντουργάνη Σταγκούλο, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Γεωργίευα, την Επίτροπο, για όλες τι ενδιαφέρουσες απόψεις τη. Ευχαριστώ και τους συναδέλφου που μίλησαν και θα ήθελα να απαντήσω σε κάποιου από αυτούς. Άκουσα και το κατά πόσον είναι κάτι το εύστοχο ή όχι το να ε, τα λέμε όλα αυτά στην Επιτροπή των Αφορών και τώρα ψάχνουμε όλα αυτά να τα ακούσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα βεβαίω να επενέσω την ε, Επιτροπή των Αφώνων γιατί νομίζω ότι εκεί προσφέρεται βήμα για τέτοιε συζητήσει και έχουμε αυτού του ε, Ευρωπαίου οι οποίοι εκεί απευθύνθηκαν. Οπότε δεν ξέρω, θα μπορούσε να ασχοληθούν και άλλε επιτροπέ, όπω η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ε, έχουμε όντω εκθέσει και άλλων ε, επιτροπών. Αλλά οι Ευρωπαίοι σε εμά έρχονται. Και όταν έρχονται όμω ζητούν απαντήσει ζητούν λύσεις στα προβλήματα. Οπότε και εμείς δεν μπορούμε τους γυρίσουμε την πλάτη. Αλλιώς δεν θα είχε νόημα η ύπαρξη της Επιτροπής των αναφορών εάν δεν ενεργούσε με τέτοιον τρόπο. θα ήθελα να πω στους συναδέλφους ότι οι αναφορές αφορούσαν την αναποτελεσματικότητα, την ανικανότητα των κρατών μελών να εκπληρώσουν τις νομικές τους δεσμεύσεις. Οπότε και εμείς προσφύγαμε σε αυτές τις αναφορές, βγαίνει από εκεί όλη αυτή η προβληματική που αναπτύξαμε και γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει αμιλητοί τα κράτη-μέλη να μεταφέρουν στο ιστορικό δίκαιο τις κοινοτικές οδηγίες και να θέσουν σε εφαρμογή τα σχετικά προγράμματα διαχείρισης απορριμμάτων και αποβλήτων. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, Ακούσαμε τι είπε και η κυρία Γεωργίβα και νομίζουμε ότι επομένω τώρα έχει προλιανθεί το έδαφος ούτως ώστε να δοκιμάσουμε για το πώς θα προχωρήσουμε προς την αυτού του προβλήματος όλες οι πολιτικές ομάδες συμφωνούν γι' αυτό και επίσης θα πρέπει να τονίσουμε το ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο απαιτεί τώρα την προσοχή μας. Χρειάζονται λύσεις από κάθε πλευρά, από κάθε χώρα Σας ευχαριστώ συναδελφοί. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση του θέματος αυτού της σημερινής διάταξης. Προσωπικά, πράγμα μου δεν θα ξανακάνω, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Είναι η πρώτη μου συνεδρία εδώ ως ε, προεδρεύοντος και συνεργαστήκατε πάρα πολύ καλά μαζί μου και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω beinahe nicht nötig zu erwähnen, aber ohne die Herren links und rechts und da. Και θέλω να πω ότι χωρίς τις κυρίες και τους κυρίους αριστερά και δεξιά από μένα δεν θα μπορούσα να είχα ε, καταφέρει τόσο καλά να ασκήσω το αξίωμα. Περνάμε όμως χωρίς καθυστέρηση, χωρίς καθυστέρηση στην έξι κυρίας